Άρχεται η συνεδρίαση. Τα κείμενα τα οποία εγκρίθηκαν στην ε, χθεσινή συνεδρίαση έχουν ε, ήδη δημοσιευθεί και ε, ρωτώ αν έχετε